το έργο. Θα ήταν επίσης ε, χρήσιμο να σκεφτόμαστε και τους ε, μισθωτούς ε, οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους πολύ συχνά κάθε μέρα επειδή οι εργοδότες τους δεν θέτουν στη διάθεσή τους τα μέσα που χρειάζεται για να προστατεύσουν τη ζωή τους στον χώρο εργασίας. Κυρίες και κύριοι, έχω να σας πιστήσω την προσοχή σε ένα σημαντικό θέμα. Ε, το προσχέδιο των, των ε, ολομελιών του επόμενου έτους ε, είναι έτοιμο. Η, σύνοση των προ... η διάσκεψη των Προέδρων συναντήθηκε στις 22 Απριλίου και οθήτησε ένα προσχέδιο ημερολογίου ε, συνόδων, το οποίο το έχετε στον χαρτοφυλάκιό σας. Στο φάκελό σας. Ε, θα το ψηφίσουμε την Τετάρτη. Και στις 18 Ιουνίου, 12 ε, το μεσημέρι, είναι η προθεσμία υποβολής ε, τροπο, αιτήσεων ε, τροπολογίας. Μιλώ για το 2011, το ημερολόγιο 2011 την Τετάρτη στις 12 θα λάβει χώρα η ψηφοφορία. Το Λαϊκό, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ε, ζήτησε ε, κάποιους διορισμούς σε, σε κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ε, έχουν, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα επιβεβαιωθούν. Κυρία Ζόλταν Μπόλτσο, Μπόλτσο και Σμιθ, μέσα Ζόλταν και Σμιθ ε, με ενημέρωσαν ότι δεδομένου ότι εξελέγησαν στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο ε, λίγη θητεία τους εδώ. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού μας και σύμφωνα με τον κανόνα 4-4 δεύτερο εδάφιο των εσωτερικών διαδικασιών μας κηρύσει τις ε, ε, θέσεις αυτές ε, χειρεύουσες από τις 14 Μαΐου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την Τετάρτη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψω 7 νομοθετικές πράξεις που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τις συνήθειες νομοθετικές διαδικασίες. Ε, οι τίτλοι αυτών των πράξεων θα δημοσιευθούν στα πρακτικά της σημερινής συνόδου. Περνάμε στην ημερήσια διάταξη. το τελικό σχέδιο ημερήσια διάταξη υιοθετήθηκε στι 12 Μαου σύμφωνα με τον κανόνα 137 και έχει διανεμηθεί. Έλαβα επιστολή από τον κύριο Κάρλο Κασίνη, πρόεδρο της Επιτροπής ε, ε, ε, Θεμάτων, που ζητάει εκ μέρους της Επιτροπής ε, η ΕΟΚΕ και η Επιτροπή των Περιφερειών να εκφέρουν γνωμοδότηση για την πρωτοβουλία των πολιτών σύμφωνα με τα άρθρα 304 ε, και 307 της Συνθήκης. Η ψηφοφορία για αυτά τα δύο ετήματα θα λάβει χώρα την Τετάρτη το μεσημέρι. Υπάρχουν σχόλια? Όχι. Περνάμε στην υιοθέτηση ημερησίας διάταξης. Δεν έχει ζητηθεί καμία αλλαγή ούτε για την ημερησία διάταξη Δευτέρα, ούτε για την ημερησία διάταξη τη τρίτη, την Τέταρτη. Τετάρτη όμως το ΕΛΚ έχει ζητήσει να συμπεριληφθεί η, ε, η έκθεση για την έκθεση Τσαρνέσκι ε, για την απαλλαγή του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κύριε Γκρέσλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί η Ισπανική Προεδρία απάντησε τα εκρεμή ερωτήματα, οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε την έκθεση και, από ό,τι φαίνεται, θα πρέπει να γίνει μια κανονική διαδικασία απαλλαγής την οποία θα συζητήσουμε με το Συμβούλιο οπότε έχουμε και τη δεύτερη σημαντική προϋπόθεση η οποία πληρείται οπότε πλέον είναι υποκοινοβουλευτικό έλεγχο το Συμβούλιο, οπότε συνιστώ εγώ στις ε, ομάδες να τεθεί αυτό το ζήτημα. Βεβαίως ε, θα το δούμε στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Σας ευχαριστώ. Υπέρ, κύριε Σπομποντα. Ναι κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομο. Συμφωνούμε με αυτό το αίτημα για τους λόγους που ακούστηκαν. Νομίζω πως θα ακολουθήσει και μια επίσημη επιστολή και ελπίζω να είναι αυτό ένα μήνυμα του Συμβουλίου πως είναι διατεθειμένο να υιοθετήσει και όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης την διαφάνεια που επέδειξε και εδώ πέρα. Οπότε συμφωνούμε με την κυρία Γκρέσλε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρος κάποιος κατά κατά αυτού του αιτήματος κύριε παρακαλώ εγώ θα έλεγα πως εκπλήσωμε εκπλήσωμε για το ότι οι δύο μεγάλες κοινοβουλευτικές ομάδες λένε να ψηφίσουμε αυτή την έκθεση εγώ ο ίδιος ήμουν σε μια συνεδρίαση των ε, συντονιστών ήρθαν πράγματι σήμερα έγγραφα από το Συμβουλίο, τα διάβασα, υπάρχει ένα παράρτημα που είναι ακριβώς το ίδιο το ίδιο παράρτημα που μας έστειλαν στις 10 Μαρτίου. Στην πράξη δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οπότε εγώ σας συνιστώ να μην τεθεί τώρα η έκθεση της στην ημερήσια διάταξη. Ειλικρινά σας λέω παίζει μαζί μας το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Θα προχωρήσουμε τώρα, πάμε στην ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ της προτάσεως του ΕΛΚ. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ. Κατά. Σας ευχαριστώ. Αποχές. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Η ψηφοφορία της εκθέσεως Τσανέσκη θα γίνει την Τετάρτη, προθεσμία υποβολής τροπολογιών. τρίτη 18 Μαΐου το μεσημέρι, στις 12 το μεσημέρι. Επίσης την Τετάρτη η ομάδα του ΕΛΚ ζήτησε η έκθεση της κυρίας Edith Bauer, Ευρωβουλευτού, για την οργάνωση του, για το ωράριο εργασίας εκείνων που ε, κινούνται στις οδικές μεταφορές να αναβληθεί ε, για την επόμενη σύνοδο, τη δεύτερη ολομέλεια. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπάουερ να αναφερθεί στο αίτημα αυτό. Στις 22 Μαρτίου η γραμματεία της Επιτροπής Απασχόλησης όταν ζήτησα να τεθεί το σημείο αυτό στην Ολομέλεια του Μαΐου μου είπαν ότι από τις 28 Απριλίου όταν θα γινόταν ψηφοφορία στην Επιτροπή μέχρι τώρα δεν ε, υπήρχε χρονικό διάστημα ενός μηνός, η περίοδος cool off και δεν μπορούσε να συμπεριφθεί το σημείο στην Ολομέλεια του Μαΐου. Χωρίς να υπάρξει διαβούλευση μαζί μου, διάσκεψη των ε, Προέδρων, πιθανότατα κατόπιν προτάσεως της σοσιαλιστική ομάδας, αποφάσισε εδώ ανεξάρτητα από το χρόνο που πέρασε να τεθεί το σημείο. Και οι πολιτικές ομάδες όμως δεν είχαν τη δυνατότητα και το χρόνο να διαμορφώσουν θέση και άποψη όσον αφορά αυτή την έκθεση. Δεν υπήρξε ο χρόνος να συζητηθεί η έκθεση και γι' αυτό εγώ ζητώ να αναβληθεί για τον Ιούνιο αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρο. Κατά να μιλήσω και ο Σφόμποντα. Κύριε Πρόεδρε, εκτιμώ την κυρία Μπάουερ, αλλά δεν ανέφερε πώς απορρίφθηκε η έκθεση. Και ξεχνάει επίσης να αναφέρει πως είναι σε επαφή με το Συμβούλιο για μια έκθεση η οποία έχει απορριφθεί. Δεν είναι αυτή η κοινοβουλευτική διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να τεθεί στην ημερήσια διάταξη. Ε, σας ευχαριστώ, λέει ο Θα ήθελα να σας πω ότι ξέχασα να ρωτήσω ποιο θέλει να μιλήσει υπέρ. κυρία Βόρτμαν Κόλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είναι μια πρόταση για την ε, νομοθετική πρόταση της Κομισιόν η οποία απορρίφθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων αλλά συνηθίζεται σε αυτό το κοινοβούλιο να έχουμε ένα μήνα μετά μία περίοδο περίσκεψης για να δούμε τι θα γίνει. Οπότε νομίζω αυτό το οποίο έκανε η εισηγήτρια είναι προς το συμφέρον του Κοινοβουλίου, είναι περίπλοκη αυτή η υπόθεση, δεν μπορούμε να το δούμε σε δύο μέρες, οπότε στηρίζω εδώ πέρα την εισηγήτρια και να το δούμε, να το ψηφίσουμε στην Ορμέλεια του Ιουνίου. Σας ευχαριστώ, θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ του αιτήματο να αναβληθεί η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Κατά. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Θα είναι η ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 158 υπέρ 137 κατά 7 αποχές οπότε γίνεται δεκτό το αίτημα. Η συζήτηση λοιπόν επί της έκθεσης Bauer αναβάλλεται για μελλοντική σύνοδο Ολομέλειας. Πέμπτη. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μας ε, ζήτησε η συζήτηση της Πέμπτης το απόγευμα για τον δημοσιογράφο στην υπερδνηστερία να αντικατασταθεί με μια συζήτηση για την κατάσταση στην Ταϊλάνδη. Οπότε αντί για την συζήτηση για τη σύλληψη του Ερνέστ Βαρντανιάν στην ε, υπερδνηστερία να συζητήσουμε την κατάσταση της ε, Ταϊλάνδης και τον λόγο έχει ο κύριος Πρέντα από αυτό. Ε, ναι, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ζήτησα να αντικατασταθεί η συζήτηση όσον αφορά την κατάσταση του δημοσιογράφου που παράνομα συνελήφθη στην υπερνιστερία και με πολύ σκοτεινές κατηγορίες να αντικατασταθεί από τη συζήτηση για την Ταϊλάνδη. Λόγω της επιδείνωσης καταστάσεως της δραματικής επιδεινούς καταστάσεως στην Ταϊλάνδη. Γι' αυτό θα θέλαμε οι συνάδελφοι όλων των πολιτικών ομάδων να εξετάσουν προσεκτικά την κατάσταση στην Ταϊλάνδη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ένας αγορητής υπέρ της προτάσεως. Θα ήθελα να ακούσω κάποιον που είναι υπέρ της προτάσεως αυτής. Ήταν μια επεξήγηση της προτάσεως αυτή που ακούστηκε. Έχετε το λόγο, ο κύριος Κασουλίδης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση στην Ταϊλάνδη χειροτερεύει ώρα με την ώρα. Ε, κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Φαίνεται ότι το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό για κατεπίγουσα συζήτηση από ότι το θέμα το οποίο θέλουμε να διαγράψουμε από, την από την ημερήσια διάξη Πέμπτης. Εν τω μεταξύ, ε, η ε, προτέτη της ε, σύλληψης του Αρνεστ Βαρντανιάν ε, έχουν προβεί σε κάποιες χειρονομίες τις οποίες θα θέλαμε να εξετάσουμε εμείς που ζητήσαμε τη συζήτηση αυτού του θέματος. Οπότε μπορούμε να δεχτούμε την αντικατάσταση. Ευχα... Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κ. Σπερώνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ό,τι και αν συζητήσουμε και αποφασίσουμε και, και την Ταϊλανδία και για την υπερνηστερία δεν αλλάζει τίποτα και γι' αυτό είναι άχρηστο να κάνουμε αναβολές να εγκρίνουμε Ε, Ευχαριστώ. Ώρα να ψηφίσουμε. Υπέρ. Ποιο είναι υπέρ τη πρόταση.